να δώσει τη γνωμοδότησή του, να σταθμεί στη θέση του από τις 17 Δεκεμβρίου 2010. Αναφέρονται λοιπόν στα πρακτικά οι τρεις αυτές προτάσει του Συμβουλίου. Τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης θα εγκριθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν δεν έχει